Ε, είπα και πριν, σε άλλους τομείς και σε άλλες πτυχές των σχέσεών μας με την Νορβηγία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος ε, που θα κλείσει τη συζήτηση, η οποία ολοκληρώνεται τώρα και αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία στις 12. Ε, Ιουλίου συνεχίζεται η συνεδρίασή μας. Έχει δημοσιευθεί η μερισσιαδιάταξη διάταξη και στην ιστοσελίδα. Κυρίσω τη λήξη των απόψινών εργασιών. Καλό βράδυ σε όλους.